αλλά δούμε αυτές τις αρχές να εφαρμόζονται και στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες του κόσμου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ συνάδελφοι των πολιτικών ομάδων που λάβετε τον λόγο και για τα σχόλιά σας και ευχαριστώ και τον Επίτροπο τον κύριο Φιούλε για τα σχόλιά του εξ της Επιτροπής. Φτάσαμε στο τέλος αυτού του σημείου της μερικής διάταξης. Περνάμε στο επόμενο. Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση η έκθεση Στάιλερ για τους εναρμονισμένους όρους εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών. Θα δώσω πρώτα απ' όλα τον λόγο στην εισηγήτρια, την Κάθριν Στάιλερ, έχει τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συνάδελφοι, είναι ωραίος τρόπος να ξεκινάμε το νέο έτος με την σημαντική αυτή έκθεση για τα προϊόντα δομικών κατασκευών και την συμφωνία που επιτύχαμε με Βιβλικής Προεδρία. Θα ήθελα λοιπόν πρώτα απ' όλα να ευχαρίσω όλους τους συναδέλφους που κατέστησαν κάτι τέτοιο δυνατό για τη σκληρή τους δουλειά, για το πώς έγινε πραγματικότητα αυτή η συμφωνία. Επίση να ευχαριστήσω την γραμματεία της επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και ιδιαίτερα τον κύριο Φερτέσεν και Χάιεκ από τη Βελγική Προεδρία για το έργο το οποίο έκαναν. Όπως λέω λοιπόν και στην εισαγωγή μου εδώ πέρα, παραφράζοντα τον ποιητή τον Ρόμπερτ ε, Φρόστ, οι καλοί φράκτε κάνουν τους καλού γείτονε. Πρέπει λοιπόν να διατηρηθεί η ορμή ολοκλήρωση τη εσωτερική αγορά και να φύγουν τα εμπόδια προς το εμπόριο. Όπως είπε και ο Μάριο Μόντι στην έκθεσή του, η Ευρώπη ακόμα είναι σε μια φασή οικοδόμησης της αγοράς κατά το οποίο απαιτεί να μην υπάρχουν εμπόριες διασυνοριακές δραστηριότητες, να μειωθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και να μειωθεί η αντίσταση των επιχειρήσεων. Με την πρόταση αυτή λοιπόν προσπαθούμε να κάνουμε την εσωτερική αγορά να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά, να έχουμε σαφέστερα συστήματα και διαφανή έτσι ώστε τα προϊόντα που ε, τίθεται στην εμπορία να είναι να πληρούν τις υψηλότερες προδιαγραφές και βεβαίω οι επιχειρήσεις να δρουν σε ένα δίκαιο περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή ο τομέα των κατασκευών αντιμετωπίζει τις οικονομικές προκλήσεις που έχει προκαλέσει η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008 και όλα αυτά επιτείνονται από την αργή οικονομική ανάκαμψη που αντιμετωπίζουμε σε ολόκληρη την Ένωση δεν πρέπει να ξεχνάμε τι σημαντικός τομέας είναι ο τομέας των κατασκευών. 12 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες απασχολούνται άμεσα και 26 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες εξαρτώνται από τον τομέα αυτόν. Μιλάμε για 38 εκατομμύρια ανθρώπους που βασίζονται σε αυτόν τον κλάδο. Για την οικονομική ανάπτυξη είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό στο τομέα των κατασκευών. Και είναι επίσης ένας πάρα πολύ επικίνδυνος τομέας. Αν δούμε τη Γερμανία που έχει τους πιο ασφαλείς κανόνες, ένας εργαζόμενος στον τομέα στου 5.000 θα υποστεί μοιραίο δυστύχημα κατά τη διάρκεια τη ζωής του. Η ασφάλεια λοιπόν όσων δουλεύουν σε αυτόν τον κλάδο σημαίνει πως πρέπει πάντα να το θυμόμαστε αυτό. Με αυτό λοιπόν κατά νου καταφέραμε και οι δύο πλευρές να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για την σήμανση επικίνδυνων ουσιών να είναι ευθυγραμμισμένο δηλαδή και με το REACH αλλά και για να δούμε τα προϊόντα εκείνα τα οποία οδήγησαν σε χρόνιες ασθένειες και θάνατο όπως παραδείγματο χάρη μεσοθυλίωμα και άντωση και Οπότε η κατάλληλη σήμανση αυτών των ουσιών μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους που έχουν τέτοιες ασθένειες των πνευμόνων. Και δείχνει αυτό πόσο σημαντικό είναι το έργο μας. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα για το ότι η έκθεση αυτή ολοκληρώθηκε το Ευρωπαϊκό Έτος του Πνεύμονα, ο οποίος συχνά παραμελείται και χαίρομαι που αναγνωρίζουμε τη σημασία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να κάνω ένα σύντομο σχόλιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πάντα λέμε πόσο ασχολούμαστε με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γι' αυτό καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ένα δεύτερο ρεύμα εμπορίας των προϊόντων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και βεβαίω θα πρέπει να είναι πιο φθηνό και πιο πρακτικό να μπορούν να το κάνουν αυτό οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κάτι το οποίο βεβαίω θα τις βοηθήσει. Για το ζήτημα της διαφάνειας και για το πώς λειτουργούν οι τεχνικοί φορείς, νομίζω πως ε, πήγαν οι φορείς έγκριση των προϊόντων περισσότερο, παραπέρα από εκεί που θα θέλαμε. Οπότε η διαφάνεια νομίζω μπορεί να ρίξει τα τείχη που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα βοηθήσει σε συνδυασμό με τις ειδικέ συνθήκες που υπάρχουν για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Και θα πρέπει βεβαίω, όπως σας είπα, να είμαστε πάντα υπέρ της καλύτερης νομοθεσίας. Εγώ, σε συνδυασμό με τους σκιοδησηγητές, συμφώνησα να διαγράψω τα κομμάτια εκείνα της έκθεσης τα οποία πλέον δεν ισχύουν. Είναι σημαντικό λοιπόν οι κανόνες να είναι σαφείς και θα ήθελα και να δω τις αλλαγές στο επιφέρει αυτή η νομοθεσία. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η κλίμακα και οι προκλήσεις, αλλά οι κανόνες αυτοί οι οποίοι θα ισχύσουν εντός 24 μηνών θα βοηθήσουν τον τομέα των κατασκευών για να δημιουργήσει ανάπτυξη και άρα θέσεις εργασίας. Ε, Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Στάιλερ, αντιπρόεδρος ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Αντώνιο Ταγιάννη έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πάνω απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο που μας κάνει την τιμή να προεδρεύει σε μια συζήτηση επί ενός θέματος τόσο σημαντικού όσον αφορά την βιομηχανική πολιτική και την πολιτική της εσωτερικής αγοράς και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Στήλε, την κυρία Στήλε, την εισηγήτρια που ε, εξέτασε εις βάθος το όλο θέμα και χάρη σε αυτή την προσπάθεια μας επέτρεψε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία στη δεύτερη ανάγνωση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πράγματι όλους τους σκιώδεις εισηγητές, τον πρόεδρο της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς, τον κύριο Χάρμπορ. Οι συνολικές συλλογικέ προσπάθειές σας ήταν αποφασιστικής σημασίας για να καταλήξουν σε μια συμφωνία μεταξύ θεσμικών οργάνων επί του άκρου τεχνικού αυτού ζητήματο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχεται θετικά το συμβιβασμό τη δεύτερη ανάγνωση από πλευρά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Και πέρα από τα τεχνικά θέματα πρέπει να πούμε ότι είναι ένα θέμα πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Η υιοθέτηση του κανονισμού για τις κατασκευές, των προϊόντων κατασκευών είναι πάρα πολύ σημαντικό βήμα για όλο τον τομέα των ευρωπαϊκών των οικοδομών τα προϊόντα των οικοδομών εκπροσωπούν το 3% του ΑΕΠ σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όσον αφορά την απασχόληση, η δραστηριότητα που συνδέεται με τις οικοδομές καλύπτουν το 6,5% του ΑΕΠ σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το 7,5% όσον αφορά ε, την απασχόληση. Άρα έχει βάρος ο τομέας των, οικοδομών της τάξης του 10% στην ευρωπαϊκή οικονομία, όπως υπενθύμησε κατά την παρέμβαση της η συγγήτρια. Η οθέτηση αυτού του κανονισμού για τα προϊόντα των, των οικοδομών είναι ένα σημαντικό βήμα πρόοδο όσον αφορά την απλούστευση και τη βελτίωση της νομοθεσίας και παγιώνει ταυτόχρονα την εσωτερική αγορά για τα προϊόντα των οικοδομών ήταν και η πρώτη υπόθεση της εφαρμογής των αρχών του Small Business Act. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες, κυρίως οι μικρότερες, επιτέλους μέσω της κοινωνικής νομοθεσίας έχουν τα κατάλληλα μέσα ούτως ώστε να μπορέσουν να ξεφύγουν από ε, το γραφειοκρατικό άχθος. Δεν μπορώ παρά να είμαι ικανοποιημένος από αυτό το αποτέλεσμα και ιδιαίτερα για τις λύσεις που δόθηκαν στα τρία ερωτήματα που ε, είχαν θεωρηθεί ε, περίπλοκα ζητήματα. Πρώτα απ' όλα το θέμα των επικινδύνων ουσιών. Εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ετοιμάσει μια έκθεση επ' αυτού του σημείου που είναι σημαντικό, ενημερώνοντας το Κοινοβούλιο και αν είναι ε, αναγκαίο θα κάνει προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου. Δεύτερον, η ειδική ε, μεταχείριση των μικρών, πολύ μικρών επιχειρήσεων, των μικροεπιχειρήσεων που θεωρούσαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές για να ε, εφαρμοστούν οι αρχές του Small Business Act. Πληρούνται τα κριτήρια βάσει του αποτελέσματο, δημιουργείται η δυνατότητα να υπάρχουν απλουστευμένε διαδικασίε για τι μικροεπιχειρήσει. Και τέλο, σε διάφορα σημεία του κειμένου αναγνωρίζεται η ανάγκη να μειωθεί το διοικητικό άκθος για τις επιχειρήσεις και για τις δοκιμές. Όχι μόνο διότι σάγονται προστευμένες διαδικασίες όσον αφορά την ετικετοθεσία για να μπει το, e, το CE, αλλά ε, για να απλουστευτούν και οι διάφορε δικασίε αξιολόγηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εξάλλου, όπω αναφέρθηκε στη δήλωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τη θέση του Συμβουλίου στην πρώτη ανάγνωση, θα πρέπει να επαληθεύσουμε ότι αυτέ οι λύσει που επελέχθησαν είναι πραγματικά οι καλύτερε για να αντιμετωπιστούν οι διάφορε ανάγκε, οι πραγματικέ ανάγκε. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να αποφύγουμε να επιβάλλουμε σε επιχειρήσει κυρίω τι πιο μικρέ από αυτέ, υποχρεώσει, διοικητικέ αδικαιολόγητε ή τουλάχιστον μη αναγκαίε. Είναι πρόθεσή μα να ελέγξουμε προσεκτικά αυτή την πτυχή και να τα εισαγάγουμε αυτά τα στοιχεία στα συμπεράσματά μα ε, που θα υποβάλουμε ε, στο Συμβούλιο και, στην, ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα πρέπει να κάνουμε μια αποτίμηση μετά από πέντε χρόνια εφαρμογή του κανονισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με το Συμβούλιο ε, για να εξετάσουμε το πώς θα εφαρμοστεί αυτός ο κανονισμός. Γι' αυτό Ζήτησα από τις υπηρεσίες μου, τις οποίες ευχαριστώ για τη συνεισφορά τους, που πάντα συνεισβάλλουν στις δραστηριότητε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζήτησα από τις υπηρεσίες να ετοιμάσουν οδικό χάρτη όσον αφορά την εφαρμογή με πρόθεσμη να σας ε, καλέσω, να σας στείλω μάλλον αυτό τον οδικό χάρτη, οπότε θα είναι έτοιμος. Λοιπόν, αναφερθώ τώρα στην επιτροπολογία. Το Κοινοβούλιο είναι ένα εταίρο πολύ βασικό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σα διαβεβαιώνω ότι προτίθεμαι να συνεχίσω τη συνεργασία στη στενή μαζί σα και όσον αφορά την επόμενη φάση που θα ακολουθηθεί μετά την οθέτηση. Ε, πέρασα 14 Πέρασα 14 χρόνια εδώ σε αυτή την αίθουσα και δεν πέρασαν εις Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προβεί σε κάποια δήλωση εν είναι αναγκαίο όσον αφορά την παρέκκληση από την κοινή συμφωνία μεταξύ των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων όσον αφορά την προθεσμία για την υποβολή ε, αντιρρήσεων όσον αφορά τι κατεξουσιοδότησης πράξη. Θέλει να υπογραμμίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η αρχή υποφασίστηκε στη στο πρόγραμμα αυτή της κοινή ε, συμφωνίας προβλέπει δύο μήνες για την προβολή αντιρρήσεων που μπορεί να παραταθεί για άλλους δύο μήνες. Σε αυτή την περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα, δεν συντρέχουν λόγοι που θα έπρεπε να δικαιολογήσουν ε, μία ε, παρέκκληση από αυτές τις αρχές. Λυπάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι η αρχή οι αρχές της κοινή συμφωνίας δεν έγιναν σεβαστές και στη δήλωσή της υπογραμμίζει ότι η περίπτωση των προϊόντων των οικοδομών δεν μπορεί να αποτελεί ένα προηγούμενο. Ε, ευχαριστώ το Κοινοβούλιο και μέσω του Προέδρου αυτού που τον ευχαριστώ για τη συμμετοχή του σε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ για τον ενδιαφέρον με το οποίο το Κοινοβούλιο εξέτασε αυτή την πρόταση απλούστευσης. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι περιμένουμε διάφορα πλεονεκτήματα από αυτή τη νέα νομοθεσία και τα αποτελέσματα που θα είναι και για τους παραγωγούς και τους χρήστες της, ε, των υλικών αυτών και για τις εθνικές διοικήσεις. Θα ωφεληθούν όλοι αυτοί. Και είναι διαθέσιμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό και να ετοιμάσει τις ε, εκθέσεις που ζητούνται. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τους αξιότιμους κυρίους βουλευτές για τη δουλειά που έκαναν και για την συνεργασία μας. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκ μέρους της ομάδας του ΕΛΚ τώρα, ο συνάδελφος Αντρέας Σφάμπ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, και εγώ θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω αυτούς οι οποίοι βοήθησαν στον πέρασε αυτός ο κανονισμός στη δεύτερη ανάγνωση. Γιατί ο κανονισμός αυτός, όπως λέει και το όνομα, επιφέρει μια βελτίωση σε σχέση με την υπάρχουσα οδηγία. Βεβαίω, το σχετικό δίκαιο αποτελούσε στο παρελθόν αυστηρά εθνική αρμοδιότητα και καταφέραμε με έναν κανονισμό της εσωτερική αγοράς να επιφέρουμε θετικέ αλλαγές. Δεύτερον, ειδικά για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. ο κανονισμό αυτό περιέχει μία σειρά σημαντικών ελαφρύνσεων, οι οποίε διευκολύνουν την κίνηση της εσωτερική αγορά. Και βεβαίω ο καταναλωτή θα ωφεληθεί όσον αφορά την ασφάλεια και την αξιοπιστία των οικοδομικών προϊόντων. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον καθηγητή τον κύριο Μάιερ και ο δισηγητή ο οποίος είναι σήμερα στην εκλογική του περιφέρεια και μου είπε να πω πως τέλος, εδώ πέρα μιλάμε για έναν καλό θετικό συμβιβασμό αλλά υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα επεξεργαστούμε περαιτέρω και ευχαριστώ τον κύριο Ταγιάννη για το ότι ανέφερε πως ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι αναμεμειγμένο και σε αυτή τη διαδικασία. Για εμάς λοιπόν δεν αρκεί μόνο να ρυθμιστεί ο παραγός και η διανομή, αλλά να υπάρχει ένα ολόκληρο πλέγμα το οποίο θα ορίζει τις αρχές και τους πρακτικούς κανόνες για τη χρήση των οικοδομικών υλικών. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την άποψη του συναδέλφου, θα πρέπει να δοθεί μια έντολη στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τυποποίησης για να βγάλει σχετικές προδιαγραφές. Τέλος, θα ήθελα να υπενθυμίσω πως η Κομισιόν θα πρέπει να παρατηρήσει εάν υπάρχει επαρκής εναρμόνιση ως αποτέλεσμα αυτού του κανονισμού και να μην οδηγηθούμε σε αθέμητο ανταγωνισμό. Είμαι λοιπόν σίγουρος, κύριε Ταγιάννη, πως θα το επιτύχουμε αυτό μαζί. Ευχαριστώ. Τώρα για την ομάδα των Σοσιαλιστών Δημοκρατών θα πάρει το λόγο η κυρία Γκέμπαχτ για δυόμιση λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κατρίν Στάιλερ, την εισηγήτρια, η οποία στο πολύ τεχνικό αυτό ζήτημα έκανε μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Γιατί δεν είναι μόνο τεχνική η έκθεση, αυτή είναι και εξόχως πολιτική. Υπάρχουν εδώ πέρα και πολιτικές που πρέπει να γίνουν σεβαστέ. γιατί το θέμα είναι να δούμε τα συμφέροντα τη οικονομία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Οπότε θα πρέπει ε, να δούμε πως είναι κάτι το οποίο το καταφέραμε εξόχως ως σοσιαλδημοκρατία. Όσον αφορά λοιπόν τα συμφέροντα της οικονομίας, είδαμε πού είναι τα προβλήματά τους στην χρήση των οικοδομικών υλικών και έπρεπε να βρεθεί ισορροπία μεταξύ των μεγάλων επιχειρήσεων και των μικρών και μεσαίων. Και σωστό ήταν αυτό το οποίο πρότεινε η Κομισιόν, δηλαδή οι μικρές επιχειρήσεις να χρειάζονται λιγότερους κανόνες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει, εξού και η βελτίωση η οποία επήλθε, δεν σημαίνει πως θα υπάρχει λιγότερη ασφάλεια και πως ε, θα ήταν χαμηλότερες οι προδιαγραφές. Και πράγματι το καταφέραμε. Βεβαίως, είναι σημαντική και η ασφάλεια. Ασφάλεια και για τους καταναλωτές η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία γιατί βεβαίως εκεί όπου χρησιμοποιείται κτίζεται ένα οικοδομικό υλικό πρέπει να φροντίσουμε ο χρήστης αυτού του προϊόντος να είναι εξίσου ασφαλής και με τον εργαζόμενο. Και τρίτον, και αυτό νομίζω είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς τους σοσιαλδημοκράτες, είναι πως έχουμε μια βελτίωση των όσων προβλέπονται για την προστασία των εργαζομένων, το οποίο γράφτηκε ακόμη μια φορά expressis verbis και έδωσε ιδιαίτερο βάρος σε αυτό η κυρία Στάιλερ, γιατί το θέμα εδώ πέρα ήταν πως έχουμε πάρα πολύ συχνά επικίνδυνες ουσίες στα δομικά υλικά και φροντίσαμε να έχουμε τον υψηλότερο δυνατό βαθμό προστασίας και αυτό έχει εξαιρετική σημασία. Και επίσης και αργότερα και πρέπει εδώ πέρα να συνεργαστούμε κύριε Ταγιάννη να δούμε τι θα γίνει με την τελική διάθεση αυτών των προϊόντων όταν δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το εξαιρετικό της έργο. Ευχαριστώ. Πολύ. Τώρα το λόγο θα πάρει η κυρία Ρούλε για την ομάδα των Πρασίνων για δύο λεπτά παρακαλώ. Äh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Στάιλερ, όλους τους σκιώδεις συγητές. Πράγματι νομίζω επιτύχαμε ένα καλό συμβιβασμό στη δεύτερη ανάγνωση, αν και πάντα πάντως συμβιβασμός δεν μπορεί να είναι όλοι ευχαριστημένοι με όλα. Οπότε θα ήθελα να αναφερθώ στις παρατηρήσεις του καθηγητού του κυρίου Μάιερ που ανέφερε ο κύριος Σφάμπ. Πιστεύω πως με τη σήμανση πρέπει να εργαστούμε περαιτέρω. Νομίζω μια καλή εναρμόνιση και της παραγωγής και των προϊόντων αυτών υπάρχει, αλλά πρέπει να δούμε και την χρήση των δομικών υλικών. Μία δυνατότητα λοιπόν είναι η Κομισιόν να εργαστεί στο πλαίσιο των Eurocodes και να τους δώσει μια σχετική εντολή. Η άλλη δυνατότητα είναι να υπάρξει μια εναρμόνιση της χρήσης για να μην ξαναπάμε στο εθνικό επίπεδο και να έχουμε μια ευρωπαϊκή μόνο στο πλαίσιο των προϊόντων και όχι στο επίπεδο της χρήσης. Οπότε και εδώ πέρα η Κομισιόν, αν θέλει να λάβει περαιτέρω μέτρα, έχει την στήριξή μας. Θα ήθελα να αναφέρω κάτι το οποίο ήταν σημαντικό στην συζήτηση και ήταν κρίσιμο για εμάς για το να συμφωνήσουμε. Υπήρχαν κάποια λάθη της Βελγικής Προεδρίας. Η Βελγική Προεδρία στη δεύτερη ανάγνωση, μετά την πρώτη ανάγνωση, εισήγαγε νέους ε, τομείς, ε, το 383 και το άρθρο 86 χωρίς την πλήρη ε, συμφωνία μας. Και βεβαίως αυτό το ανέφερε η Ουγγρική Προεδρία σε μια επιστολή της. Δεν νομίζω βεβαίως να είχε αντιληφθεί πλήρως εδώ πέρα την σύγκρουση. Θα ήθελα να υπενθυμίσω πως προσεχώς ε, όταν θα φέρνει νέα σημεία στη δεύτερη ανάγνωση στο Συμβούλιο θα είναι υποχρεωμένο να έρχεται πιο πολύ προς την μεριά του Κοινοβουλίου. Οπότε Βεβαίω συμφωνούμε πως δεν έχει νόημα να καταψηφίσουμε την έκθεση λόγω ενός πραγματικά τυπικού λάθους. Συμφωνούμε λοιπόν, χρειάζεται εναρμόνιση ο κλάδος και έχει πάρα πολύ μεγάλη οικονομική σημασία. Γι' αυτό λοιπόν, όπως σας είπα, υπερψηφίζουμε στη δεύτερη ανάγνωση. Και τώρα το λόγο θα πάρει για τους συντηρητικούς μεταρρυθμιστές η κυρία Μακ Λάκριν για ένα λεπτό παρακαλώ. Ε, σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Στάιλερ για τη σκληρή δουλειά ήταν πολύ μακρύς ο δρόμος. Σήμερα στην Ευρώπη ο τομέας της οικοδομής ε, απασχολεί 12 εκατομμύρια περίπου πολίτες και το 90 περίπου της 100 των, ε, κατα... των κατασκευαστών δομικών υλικών είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 65.000 δηλαδή μεμονωμένες επιχειρήσεις. Άρα ο τομέας της οικοδομή είναι ζωτική σημασία ε, για την ευρωπαϊκή οικονομία. Έχουμε ευθύνη απέναντι στον κλάδο. Ιδίω μετά την οικονομική κρίση πρέπει να τον στηρίξουμε. Υπάρχει ίσως ε, ένα πρόβλημα, υπάρχει ε, ένα πρόβλημα με το με την νομοθεσία. Δεν είναι τέλεια, αλλά είναι ένα συμβιβασμό. Υπάρχουν σημαντικά ε, σημεία τα οποία υπάρχουν. Δήλωση απόδοση, σήμανση CE. Θέλουμε να μην υπάρχει ο ίδιο φόρτο για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Θα πρέπει επίση να επισημανθούν και να εντοπιστούν επικίνδυνε ουσίε. Εδώ υπήρξε συνένεση για να μην έχουμε και ε, αντίφαση και σύγκρουση με ήδη υφιστάμενε νομοθεσίε. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την ελεύθερη κυκλοφορία δομικών υλικών, να βελτιώσουμε τα πρότυπα ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση και να προωθήσουμε και την ανακύκλωσή του στο μέλλον. Κυρίω όμω να μην αυξήσουμε το γραφειοκρατικό άκτο ούτε των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ούτε των καταναλωτών. Τώρα ερχόμαστε στον κατάλογο των άλλων εγγεγραμμένων μιλητών. Η κυρία Κόμη για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, χαιρετίζω τον επιτεθέντα συμβιβασμό και αναφορά σε διάφορα σημεία τα οποία θεωρώ ότι είναι ζωτική σημασία σε αυτά που υπογραμμίζονται. Ανεπαρκή εφαρμογή των στόχων, υλοποίηση των στόχων που με τέτοια νομοθετική πρόταση προτείνουμε να επιτευχθούν. Αναφέρομαι στη διατήρηση των προδιαγραφών όσον αφορά τι απλουστευμένε διαδικασίε θα πρέπει να ελαφρύνουμε το άχθος και να μειώσουμε το κόστος για τις επιχειρήσεις. Πολύ συχνά όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι μεγάλο το βάρος. Είναι απαραίτητο πιστεύω στα πλαίσια μιας οικονομικής συγκυρίας που είναι αρνητική όπως είναι η παρούσα να γνωρίζουμε τη σημασία του ρόλου που παίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να αναγνωρίζετε. Είναι ένας βασικούς πυλώνες επί των οποίων βασίζεται η οικονομία μας, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πέραν αυτού, μέσω μηχανισμών διαδικαστικών που είναι απλουστευμένοι και πιο συγκεκριμένα με την μείωση του χρόνου για την διάθεση νέων προϊόντων στην αγορά, η νέα νομοθεσία ευνοεί την κοινοτομία. Ταυτόχρονα προστατεύει τους καταναλωτές δημιουργώντας τις συνθήκες για να μπορούν πιο έγκαιρα να ε, χρησιμοποιούν αυτά τα προϊόντα χωρίς να παρατηρούνται από τις εγγύσεις που υπάρχουν την ασφάλεια και την εγγύηση που θα πρέπει από το σήμα CE να ξέρουν ότι είναι εγγυημένα. Η επιτευχή σας συμφωνία κατά την αποψή μου είναι έξοχο συμβιβασμό που μπορεί να πετύχει τη σωστή εξισορρόπηση μεταξύ απαιτήσεων των παραγωγών και απαιτήσεων των καταναλωτών και εγγυάται έτσι τη σωστή λειτουργία της αγοράς σε έναν τομέα που είναι πραγματικά πολύ βασικός για την οικονομία την ευρωπαϊκή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Η κυρία Ράπτη για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Όπως ευχαριστώ πάρα πολύ και την Κάθριν Στάιλερ για την εξαιρετική δουλειά που έκανε. Μιλήσαμε όλοι για ένα τεχνικό θέμα και ευτυχώς η κυρία Γκέπχαρτ εκ μέρους των Σοσιαλιστών υπογράμμισε ότι δεν είναι μόνο τεχνικό θέμα. Είναι ένα άκρος πολιτικό και οικονομικό θέμα. Η οικοδομή ξέρουμε όλοι ότι είναι βασικός πυλώνας της οικονομίας οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ξέρουμε όλοι ότι είναι η σπονδυλική στήλη της οικονομίας μας μιας οικονομίας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ένωσης που βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. άρα λοιπόν η έκθεση της κατρίν είχε μια έντονη πολιτική σημασία και τα κατάφερε περίφημα. καταφέραμε και είχαμε ένα συμβιβασμό ένα καλό συμβιβασμό για όλους καταφέραμε να βρούμε την ισορροπία εκείνη που θα μας δώσει απλές διαδικασίες τις οποίες θα μπορούν να εφαρμόσουν χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ταυτοχρόνως το μέγιστο δυνατό καλό αποτέλεσμα. καταφέραμε να χτυπήσουμε την υπόθεση των επικίνδυνων ουσιών όλοι θυμόμαστε και οι παλαιότεροι μου εδώ πάρα πολύ καλά την υπόθεση της μόλυνσης με τον αμίαντο του κτηρίου του μπερλεμόντ που είχε κλείσει για πέντε ή έξι χρόνια. για φανταστείτε τι θα γίνει σε ολόκληρες πολιτείες μέσα στην ευρωπαϊκή ένωση εάν δεν θα μπορούσαμε να χειριστούμε το θέμα των επικίνδυνων ουσιών έχουμε τέλος μπροστά μας ακόμη το θέμα της ασφάλειας και της διαφάνειας και εδώ νομίζω ότι τα κατάφερε περίφημα η κατρίν στην έκθεσή της και στο συμβιβασμό που επιτεύχθηκε. κλείνοντας κυρία πρόεδρε και σας ευχαριστώ για την ανοχή θα ήθελα να ευχηθώ τόσο καλά όσο καλά τα καταφέραμε στην οικοδομή άλλο τόσο καλά να μπορέσουμε να, τα καταφέρουμε στην οικοδόμηση της ευρωπαϊκής πολιτείας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ράπτη. Ο κύριος Χάρμπουρ θα πάρει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ως Πρόεδρος Επιτροπής Θέλω να συμφωνήσω με πολλές ή μάλλον με όλες τις παρατηρήσεις που άκουσα για τη δουλειά που έχει κάνει η Κάθριν Στάιλερ αναλαμβάνοντας ένα πολύ πολύπλοκο θέμα για τη δεύτερη ανάγνωση ε, πραγματικά επιτέλεσε αξιοθαύμαστα το πολύ δύσκολο καθήκον που ανέλαβε. Βλέπουμε κυρία Πρόεδρε τη σημασία που έχει τελικά η διαδικασία της δεύτερης ανάγνωσης ε, στο σώμα αυτό. Διότι καταφέραμε να ε, βελτιώσουμε σημαντικά το κείμενο το οποίο είχαμε παραλάβει, δηλαδή την κοινή θέση, την κοινή θέση του Συμβουλίου. Όπως επισήμανε ιδιαίτερα η κυρία Ρούλε υπήρξαν διαφωνίες, λάβαμε και επιστολή από την Ουγγρική Προεδρία, θα δημοσιευθεί μαζί με τα πρακτικά για κάποια από τα πιο αναλυτικά ζητήματα. Θα ήθελα να κάνω δύο καταληκτικές παρατηρήσεις ε, και να εκφράσω βέβαια και τη συμφωνία μου με την ε, θέση αυτή. Πρώτα απ' όλα να πω ε, στον Επίτροπο. Σας ευχαριστώ που συνεργαστήκατε μαζί μας. Πρέπει να συνεργαστούμε και στενά σε ό,τι αφορά την εφαρμογή. Είπατε κι εσείς ότι υπάρχουν σημαντικές πτυχές ε, που έχουν να κάνουν με τη διαδικασία της Επιτροπής. Η δική μου επιτροπή πιστεύει πραγματικά ότι θα πρέπει να παρακολουθήσουμε πάρα πολύ προσεκτικά τις προτάσεις αυτές και την εφαρμογή τους. Δεύτερον, είναι ένας τομέας κρίσιμο, ζωτική σημασία. Είπαν και προλαλήσαντες ότι πρέπει να φροντίσουμε να μην υπάρξουν φραγμοί, να μην υψωθούν εμπόδια που να ε, εμποδίσουν τον τομέα αυτό να συμβάλλει όσο το πράττει μέχρι σήμερα στον τομέα. Είναι ομιλήτρια η κυρία Κορχόλα, δεν φαίνεται να είναι στην αίθουσα, οπότε ερχόμαστε κατευθείαν στη διαδικασία Catch the Eye. Έχουν ζητήσει δύο συνάδελφοι να παρέμβουν. Ε, θα πάρουν το λόγο από ένα λεπτό. Η κυρία Ρότοβα, παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το θέμα αυτό το έχουν παρακολουθήσει οι επίτροποι Ταγιάννη και Μπαρνιέ. Θα πρέπει να έχουμε νέα σήμανση, τεκμηρίωση, ε, να εξαλειφθούν οι αχρίαστες γραφειοκρατικές πρακτικές στον τομέα των δομικών υλικών. Πρέπει να παρέχουμε κατασκευαστικές υπηρεσίες σωστές. Όλες ε, οι υπηρεσίες πιστεύω ότι θα εκτιμήσουν τις μεταρρυθμίσεις αυτές ιδίως στην Τσεχία. Συμπεριλήφθη, αναφορά και τι πολύ μικρέ επιχειρήσει. Στην Επιτροπή μα υπήρξε συμφωνία. Ελπίζω και στην Ολομέλεια και στην ψηφοφορία να υπάρξει ομοφωνία για να στηρίξουμε και την ενιαία αγορά. Ευχαριστώ κύριε Ροϊτοβά. Τώρα το λόγο θα πάρει η κυρία Βέσ Γκέρμπερ. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν έχω πιστεί σε όλα τα σημεία, αλλά αναγνωρίζω πως πρόκειται για μια σαφή βελτίωση σε σχέση με την υπάρχουσα κατάσταση, γιατί για πρώτη φορά έχουμε ενιαία ευρωπαϊκή τεχνική γλώσσα για τις επιδόσεις των οικοδομικών υλικών και απλοποιημένες διαδικασίες και αυστηροποιημένες διαδικασίες. Οπότε προωθήσαμε έτσι την ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά και τις ε, εταιρείε αλλά και μέσω των αυξημένων απαιτήσεων ασφαλείας βοηθήσαμε και τους καταναλωτέ. Επίσης, σημαντικό είναι αυτό το οποίο έγινε, δηλαδή η μείωση τη γραφειοκρατία για τις μικρομισέ επιχειρήσει, αλλά θα πρέπει να δούμε πως μεταξύ των χρηστών είναι και μικρομισές επιχειρήσει, οι οποίες επίσης προστατεύονται. Οπότε χαίρομαι για το ότι η πρότασή μου έγινε δεκτή δηλαδή να ισχύσουν απλοποιημένες ε, διαδικασίες για τις πολύ, μικρόμεσες, για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις χωρίς αυτό να σημαίνει πως είναι λιγότερο αυστηρές. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε αξιόπιστες ενδείξεις, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ασφάλεια των κτηρίων σε όλο την Ευρώπη. Ευχαριστώ. για το θέμα αυτό. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, οπότε το λόγο θα πάρει ο Επίτροπος, ο κύριος Σταγιάννη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. με τα λόγια του Προέδρου, του κύριου Άρμπορ, που υπογράμμισε τη σημασία του κειμένου που συζητούμε, το οποίο θα εγκριθεί χάρη σε αυτή τη συμφωνία, θα εγκριθεί από την Ολομέλεια, διότι πρόκειται περί νέου κανονισμού, νέας νομοθεσίας που θα στείλει μηνύματα σημαντικά προς την αγορά αλλά ταυτόχρονα θα καθορίσει καλούς κανόνες, σωστούς κανόνες που θα επιτρέπουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορούν να αναπτυχθούν. Κυρίως σε αυτή τη φάση, την τελική φάση της κρίσεως όπου εμείς πρέπει να κάνουμε τα πάντα, ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορούν να δημιουργήσουν νέα απασχόληση και να μπορούν να αναπτυχθούν. Αυτός είναι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που το είδαμε και το συμμερίζεται και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις προσπάθειες που κατέβαλε χάρη και στην εφαρμογή και ανάπτυξη του Small Business Act. Απλούστευση λοιπόν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, άρα μείωση των γραφειοκρατικών βαρών αλλά θεσπίζοντας τους κανόνες για την ε, απελευθέρωση της αγοράς, για την ανάπτυξη της αγοράς, όπως είπε και η κυρία Γκέπαρτ, είναι ένα μήνυμα αυτό που στέλνουμε, που αφορά και την ασφάλεια. Την ασφάλεια που έχει μεγάλη σημασία για τους εργαζομένους του τομέα, των κατασκευών και των οικοδομών και για τους καταναλωτές. Και θεωρώ ότι αυτό το κείμενο ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση. Βέβαια, με την επιφύλαξη ότι είναι πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μην ολοκληρώσει προσπάθειες με την έγκριση των προδιαγραφών αυτών της νομοθεσίας που είναι καρπός του συμβιβασμού μεταξύ Συμβουλίου και, και Κοινοβουλίου. Θέλουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε τα επόμενα χρόνια και το, σας διαβεβαιώνω, επίσημα αναλαμβάνω αυτή τη δέσμευση, το υπογράφησε ο κ. Χάρμπορ. Πρέπει να προχωρήσουμε, να δι... καταρτήσουμε έναν οδικό χάρτη όσον αφορά την εκτέλεση αυτών των μέτρων που θα σας αποστείλω όποτε θα είναι έτοιμος, όποτε θα είναι δυνατόν. Πολλοί βουλευτές κατά τη διάρκεια της συζητήσεως μίλησαν αναφερόμενοι στο θέμα της εναρμόνισης στον τομέα των ε, κατασκευών κυρίως όσον αφορά την ασφάλεια. Έχω πλήρη επίγνωση. Ξέρω το πρόβλημα και χαίρομαι που έχουμε ετοιμάσει τους, ε, τις προδιαγραφές ευρωπαϊκές, τις αναρμονισμένες προδιαγραφές που αφορούν ε, την ασφάλεια των οικοδομών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως γνωρίζετε, αυτή τη στιγμή ετοιμάζει μια ανακοίνωση όσον αφορά το θέμα της τυποποίησεως ε, που θα υποβληθεί ε, σε μερικές εβδομάδες και θα τεθεί στην προσοχή του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, πιστεύω ότι σήμερα και αύριο πραγματοποιείται ένα σημαντικό βήμα προόδου. Επαναλαμβάνω, δεν πρόκειται μόνο και ευχαριστώ για την υπομονή της εισηγήτριας που ετοίμασε, που αναφέρθηκε στις τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν μια φωτογράφηση των πολιτικών δεσμεύσεων που αναλύθησαν. Είναι προδιαγραφές που δεν είναι απλώς τεχνικές, πίσω από τη τεχνικά χαρακτηριστικά κρύβεται μια επιλογή οικονομική, σημαντική επιλογή. Το επαναλαμβάνω. Υπέρ των μικρομεσών επιχειρήσεων, που εκείνε οι επιχειρήσει μπορούν να δημιουργήσουν νέες θέσει τα επόμενα χρόνια. Και είναι η υπέρ των, των 500 εκατομμυρίων ε, Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, και τη συζήτηση θα κλείσει η συγγήτρια η κυρία Στάλερ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους ε, οι οποίοι μίλησαν ε, απόψε για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι ο κύριος Ταγιάννη, το σχόλιο του κύριου Ταγιάννη για την εταιρική σχέση και για τον οδικό χάρτη και σε σχέση και με αυτό που είπαν οι κύριοι Σφάπ κυρία, ο κύριος Σφάπ και η κυρία Ρούλη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή πρέπει να συνεχίσουμε την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε. Φτάσαμε σε ένα συμβιβασμό, ίσως υπήρχαν κάποια ε, πράγματα που ήθελαν κάποιοι συνάδελφοι να συμπεριληφθούν δεν συμπεριελήφθησαν. Το 75% όμως των τροπολιών που εμείς θεωρούσαμε σημαντικές έχουν γίνει δεκτές και ε, αυτό είναι θετικό. Είναι πάρα πολύ ζωτική σημασία για τι οικονομίε μα, για τη μελλοντική ανάπτυξη τη θέση εργασία, ο τομέα τη οικοδομή, ο τομέα των κατασκευών. Θέλω λοιπόν να, να ρωτήσω τον κύριο Αντιπρόεδρο, θα μπορούσαμε μήπω να έχουμε, και μάλιστα την κυρία Αντιπρόεδρο συγκεκριμένα, να έχουμε μια ετήσια συζήτηση για αυτά τα ζητήματα ε, στο κοινοβούλιο ώστε πάντοτε να βάζουμε ε, στο επίκεντρο, να δείχνουμε την πραγματική σημασία που έχει ο τομέα τη οικοδομή. Είναι εκατομμύρια οι πολίτε που βασίζονται για τι θέσει, για δουλειέ του στον τομέα αυτό. Σα ευχαριστώ λοιπόν κύριε Επίτροπε και πραγματικά προσβλέπω σε επόμενου μήνε και έτη θα έλεγα γιατί φαντάζομαι ότι θα συνεχιστεί και στην Επιτροπή Ιστορική Αγορά η συζήτηση για το τομέα τη οικοδομή και εμεί θα τον παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ. Ευχαριστώ κυρία Στήλε απευθύνατε και προτάσεις στο Προεδρείο, τις οποίες σημειώσαμε. Η διάσκεψη των Προέδρων μπορεί να ε, το συζητήσει και να έχει μια απάντηση για το θέμα σας.